Ε, Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού μας, και βάσει άλλων στοιχείων του κανονισμού κοινοβουλευτικής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω να κάνω μια ανακοίνωση σε εσάς που απαριθμεί τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προεδρού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού δεν θα υπάρξουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. Έχω λάβει τις εξής προτάσεις υποψηφιότητος για τον, το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Νέρτς Ντίβα, καταρχήν. Αν μπορείτε να σταθείτε όρθιος αγαπητές συνάδελφε. Μάρτιν Σούλτς και η κυρία Νταϊάννα Γόλης είναι οι τρεις υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου. Με έχουν πληροφορήσει οι τρεις υποψήφοι ότι συμφωνούν με την πρόταση υποψηφιότητός τους. η, η σύνθεση του Κοινοβουλίου σήμερα θα εμφανιστεί στα πρακτικά και κλείνουμε έτσι τη συνεδρίασή μας σήμερα. Σας ευχαριστώ και θα βρεθούμε αύριο για την ψηφοφορία.